μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πάντοτε υποστήριξα τη φιλευρωπαϊκή στάση. Μετά από 9 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου δεν δημιούργησα κανένα σκάνδαλο, όπως εσείς δεν έκανα καμία σκηνή, ε, όπου συμφώνησα με όλες τις θετικές λύσεις για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν μπορώ να τοποθετηθώ τώρα κατά αυτών των ε, θεσμικών οργάνων. Ε, εγώ άσκησα κριτική στο ψήφισμα γιατί πίστευα και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε αυτήν την ενότητα. Μιλήσατε για τις διαδηλώσεις ε, της 10ης Αυγούστου στη Ρουμανία. Τι λέτε για τις διαδηλώσεις στη Γαλλία. Ποια στάση έχετε εσείς. Εγώ δεν θέλω να αναφερθώ στο θέμα αυτό γιατί η Γαλλία λαμβάνει τις δικές της αποφάσεις. Όμως, ούτε κανένας, ούτε κάποιος Γάλλος βουλευτής, ούτε κανένας Ευρωπαίος βουλευτής ήρθε εδώ για να επικρίνει τη χώρα του, τη Γαλλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και πιστεύω ότι η δική μας στάση μετρά για τους πολίτες που μας βλέπουν από το σπίτι τους. Κάνατε μια πολύ σοβαρή δήλωση σε σχέση με την ελευθεροτυπία. Σας διαβεβαιώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, διαβεβαιώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η κυβέρνηση της Ρουμανίας δεν έχει καμία σχέση με κάτι τέτοιο. Αυτό σημαίνει παραπληροφόρηση. Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Πράγματι, ένα τηλεοπτικό κανάλι είδε να διακόπτεται την εκπομπή του για 10 λεπτά. Αυτό αποφασίστηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος. Η ρουμανική κυβέρνηση δεν έχει καμία σχέση με αυτό το ζήτημα. Όμως, ταυτόχρονα, θα πρέπει να δούμε για να δώσουμε περισσότερη αξιοπιστία στις δικές μας αποφάσεις, να είμαστε προσεκτικοί στις δηλώσεις που κάνουμε. Και αυτά που λέμε να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, γιατί διαφορετικά όλοι μας θα κριθούμε. Όμως το πιο σημαντικό είναι ότι θα κριθεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που χρήζει ενός καλού μέλλοντος. Σας ευχαριστώ και πάλι βασίζομαι στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην διαδρομή μας. Σας ευχαριστώ. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε και τώρα η μερίσια διάταξη προβλέπει την έκθεση του κυρίου Μάτο ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2017. Κύριε Γιούρεκ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρέπει να πω για τον κύριο Μπούλμαν ότι ε, θέλω να ζητήσω το λόγο για ένα διαδικαστικό. Το να έχει κανεί δικαίωμα να λάβει το λόγο είναι κάτι που προβλέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου. Δεν είναι προνόμιο. Ε, πέραν αυτού και σύμφωνα με το σχετικό άρθρο του εσωτερικού κανονισμού, είναι πολύ σαφέ για το ποιος ε, πώ θεμελιώνεται το δικαίωμα αυτό και τι δικαίωμα έχει ο πρόεδρο τη Ολομέλεια να κρίνει και να αποτιμά τον κανονισμό αυτό, δίνοντα το λόγο στου μεν και στου δε. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδε να χρησιμοποιείται ο όρος φασίστας εδώ για μέλη ή κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν μπόρεσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω, κύριε Σασόλη. Ε, όταν προέδρευε ο κύριος Σασόλη μάλλον. Και ε, εδώ ήθελα να παρέμβω στη συζήτηση αυτή. Δεν μπορούμε να συμπεριφερόμαστε στο Κοινοβούλιο κατά τον τρόπο αυτό. Ε, πρόκειται για μια από τις υποχρεώσεις του Προέδρου της Ολομέλειας να παρέχει δικαίωμα παρέμβασης στον καθένα από τους ευρωβουλευτές. Πολλές φορές μιλάμε για ανελεύθερα δημοκρατικά καθεστώτα και για να μπορούμε κι εμεί να υπερηφανευόμαστε για τη δημοκρατία μα εντό του κράτου δικαίου, θα πρέπει να έχουμε εμεί πρώτη υποδειγματική συμπεριφορά, εδώ μάλιστα, στην ε, Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Μάλιστα, θα φροντίσω να, ακούσω το απόσπασμα για να δω τι ακριβώς συνέβη και θα τοποθετηθώ μετά. Attendiamo Draghi. Περιμένουμε τον πρόεδρο Ντράγκη. Ο κύριος εισηγητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε, κύριε Ντράγκη. Πάντοτε είναι ικανοποίησή μα να σα έχουμε εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα τους σκιώδει εισηγητέ και όλου του συναδέλφου για τη μεγάλη υποστήριξή του και τη συνεργασία, ώστε να μπορέσω να παρουσιάσω μια καλή έκθεση το ευρώ συμπληρώσει 20 έτη και είναι σε μια στιγμή που είναι πιο δημοφιλέ. Τρει στου τέσσερι πολίτε πιστεύουν ότι ωφελεί την οικονομία μα. Αυτό που ξεκίνησε ω κοινό νόμισμα για 11 χώρε, σήμερα είναι για 19 και 340 εκατομμύρια κατοίκους. Επιπρόσθετα, το ευρώ γιορτάζει την 20η επαιτειό του μετά από ένα μεγάλο έτος το 2017. Η ευρωπαϊκή οικονομία μεγενθήθηκε με το πιο ισχυρό ρυθμό της τελευταίας δεκαετίας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα κράτη-μέλη είδαν ότι μεγενθήθηκαν οι οικονομίες τους και πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτό οφείλεται τόσο στην νομισματική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, όπω και στι διορθωτικέ μεταρρυθμίσει ε, που υλοποίησαν πολλά κρατημέλη. Τα τελευταία δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από τη Eurostat πέρσι τον Ιούλιο μας δείχνουν ότι πηγαίνουμε στην ορθή κατεύθυνση. Η οικονομική μεγένθηση για το 2018 και 2019 παγιώνεται στο πάνω από 2%. Η ανεργία τοποθετείται βασικά σε ε, επίπεδα προκρίσεις γύρω στο 7% και ταυτόχρονα ο αριθμός των απασχολούμενων και η αναλογία της συμμετοχής στην αγορά εργασίας της Ευρωζώνης βρίσκεται στο πιο υψηλό επίπεδο από την δημιουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης το 1999. Όμως δεν είναι όλα θετικά. Ε, με ανησυχεί η έλλειψη σύγκλησης και η τάση κάποιων κρατών μελών να μην ε, αντιμετωπίζουν τα διεθνωτικά τους ελλείμματα. Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό, η ΕΕΚΤ, της οποίας η ανεξαρτησία είναι θεμελιώδης, ε, υλοποιεί την εντολή της να διατηρήσει τον πληθωρισμό κάτω αλλά γύρω στο 2%. Μεσοπρόθεσμα αναμένεται ότι το 2018, 19 και 20 ο πληθωρισμός θα είναι γύρω στο 1,7% και αυτό σίγουρα οφείλεται στα μέτρα που υιοθετήθηκαν. Επίση, είδαμε βελτίωση τη χορήγηση πίστος στο ιδιωτικό τομέα το 2018, αυξήθηκε με ένα αριθμό 3% ετησίω. Λεχθέντω αυτού, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, επειδή προκύπτουν βεβαιότητε γύρω από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανάδυση του λαϊκισμού και τις πιθανές συνέπειες ε, του Brexit και τον προστατευτισμό μεταξύ άλλων πολλών κινδύνων. Θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο ουσιαστικό, δηλαδή να εγγυηθούμε ότι συνεχίζουμε στην κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θεσίων εργασίας. Ε, αυτή είναι η πραγματική κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό είναι ζωτικό να διατηρήσουμε ένα ευνοϊκό σενάριο για ιδιωτικέ και δημόσιε επενδύσει και να φτάσουμε σε επίπεδα προκρίση. Προ την πτυχή αυτή, χρειάζεται μεγαλύτερη δράση από την πλευρά τη ΕΚΤ για να εγγυθεί ότι η νομισματική τη πολιτική θα πετύχει το στόχο να ξαναδώσει κονδύλια στην πραγματική οικονομία, κυρίως στη ΜΜΕ, που είναι η σπονδυλική στήλη της οικονομίας μας και τα μέτρα νομισματικής επέκτασης να ωφελήσουν την κοινωνία στο σύνολό τη. Στην έκθεση που προετοιμάσουμε και θα ψηφίσουμε αύριο, έχουμε συμπεριλάβει όλες τις στοιχείες που αναφέρονται στην νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αξιολογώντας τα μέτρα που έπρεπε να υιοθετηθούν, αλλά καλωσορίζοντας και την απόφαση προαιρευτικής μείωσης αυτών των μέτρων ε, όταν το επιτρέπει η οικονομική κατάσταση και ε, εδώ τονίζουμε την ε, μείωση του προγράμματος περιουσιακών στοιχείων, ε, την έναρξη του προγράμματος εταιρικών ομολογιών και το πρόγραμμα της αγοράς δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη μεταξύ άλλων. Η ΕΚΤ δεν μπορεί να επιλύσει τα διορθωτικά προβλήματα των κρατών μελών. Είναι τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα που πρέπει να δράσουν σε εθνικό επίπεδο για να δημιουργήσουν υγιή θεμέλια πάνω στα οποία θα βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα μέτρα τη ΕΚΤ έχουν μεταβατικό χαρακτήρα και το κύριο πλεονέκτημά του είναι ότι δίνουν χρόνο στα κράτη-μέλη έτσι ώστε αυτά να μπορέσουν να εξηγιάνουν την δημοσιονομική του κατάσταση και να εφαρμόσουν διαφορετικέ μεταρρυθμίσει που θα δημιουργήσουν τι προποθέσει για να συνεχίσουν στην οδό τη οικονομική ανάπτυξη. Και όλοι ενεχόμαστε σε αυτό. Σα ευχαριστώ. Τον λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο κύριος Μάριο Ντράγκη, τον οποίο ευχαριστώ που δέχτηκε την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να έρθει στις ε, πανηγυρικές εκδηλώσεις για τα 20 χρόνια του ευρώ και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα για να συζητήσουμε τις δραστηριότητες της ΕΚΤ και το σχέδιο ψηφίσματός σας για την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2017, πριν από 20 χρόνια. Την 1η Πρώτου 1999 ε, εισήχθη επισήμως το ευρώ και ξεκίνησε το ευρωσύστημα τις ε, νομισματικές του δραστηριότητες ε, και είχαμε μια κοινή νομισματική ζώνη 11 χωρών. Ένα ιστορικό βήμα για την ε, Ήπειρό μας και οπωσδήποτε ένα άλμα προς τα εμπρός στην οικονομική μας ολοκληρώση. Η 20η επέτειος μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια ανασκόπηση στις επιτυχίες που είχαμε αλλά να σκεφτούμε και το τι ακόμα πρέπει να γίνει έτσι ώστε το ευρώ να αποδώσει πλήρως. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα επί τη ευκαιρία να κάνω μια ανασκόπηση στην νομισματική πολιτική της ΕΚΤ για να δούμε το τι διδαχτήκαμε και να τονίσουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Θα εστιάσω κυρίως τα τελευταία 7 χρόνια τα οποία συμπίπτουν με την δική μου θητεία οι δύο δεκαετίες ύπαρξης ε, του ευρώ ε, πραγματικά είναι πάρα πολύ διαφορετικές. Η πρώτη ήταν το αποκορύφωμα μιας ε, τριακονταετίους περίοδους μακροοικονομικής σταθερότητας. Η δεύτερη δεκαετία μετά είχε την χειρότερη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση από τη μεγάλη ύφεση. Βεβαίως, φυσικό είναι, οι δύο αυτές ε, περίοδοι να απαιτούν διαφορετική νομισματική πολιτική και διαφορετικά εργαλεία για να εφαρμοστεί αυτή. Η περίοδος πρώτης ε, κρίσης ε, είχε μικρές μεταβολές στον οικονομικό κύκλο και έτσι η ΕΚΤ μπορούσε να διασφαλίσει σταθερότητα των τιμών κυρίως μέσω των επιτοκίων. Όμως η κρίση του 2008 άλλαξε θεμελιωδώς το οικονομικό τοπίο εντός του οποίου λειτουργούμε. Νέα μέσα απαιτήθηκαν για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής και να σταθεροποιήσουμε την οικονομία της Ευρωζώνης. Αυτό με τη σειρά του απέτησε να αλλάξουμε προσέγγιση όσον αφορά την επικοινωνία και την λογοδοσία της Κεντρικής Τράπεζας. Όταν ανέλαβα καθήκοντα τον Νοέμβριο του 2011 η Ευρωζώνη αντιμετώπιζε πολύ δύσκολες συνθήκες. Η οικονομία είχε ανακάμψει από την κρίση της Λίμαν ε, με τρόπο παρόμοιο όπως και άλλες νομισματικές ζώνες. Αλλά από το 2010 και μετά είχαμε μια απώλεια εμπιστοσύνη στην βιωσιμότητα του κρατικού χρέους και αυτό δημιουργούσε έναν φαύλο κύκλο αυξανόμενου κόστους δανεισμού, κατακαιρματισμού και μειούμενης οικονομικής δραστηριότητας. Οι περικοπές ε, και στα επιτόκια της ΕΚΤ δεν περνούσαν ε, στις επιχειρήσεις ε, και στα νοικοκυριά στον ίδιο βαθμό σε κάθε χώρα της Ευρωζώνης. Υπήρχε λοιπόν μια δυσλειτουργία του μηχανισμού νομισματικής μετάδοσης, την οποία ναι, αν δεν φροντίζαμε θα είχαμε ένα πρόβλημα για τη σταθερότητα των τιμών. Η ΕΚΤ αντέδρασε με δύο πολιτικές. Πρώτα απ' όλα υπήρχε ε, ρευστότητα από τις κεντρικές τράπεζες στις τράπεζες για μέχρι και τρία χρόνια και υπήρχαν διάφορα στοιχεία ως εγγυήσεις ε, η φύση των οποίων επεκτάθηκε. Έτσι μειώθηκε ο κατακαιρματισμός της συνθήκης χρηματοδότησης των τραπεζών. Και δεύτερον, η ΕΚΤ ανακοίνωσε αυτό το οποίο λέμε outright monetary transactions, τις νομισματικές συναλλαγές, το 2012, κάτι το οποίο πλέον σήμαινε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος αλλαγής νομίσματος όσον αφορά τα κρατικά ομόλογα. Όμως ε, αυτή η κρίση άφησε βαθιά σημάδια στην οικονομία. Ανέβηκε πολύ η ανεργία, οι, επεν... οι εταιρείε μείωσαν τις επενδύσεις και η μη εξυπηρέτηση των δανείων αυξήθηκε. Παρά το ότι μειώθηκε ο δημοσιονομικός κατακαιρματισμός, οι τράπεζες άρχισαν να μειώνουν τους ισολογισμούς τους και δεν ήθελαν να δανείζουν. Έτσι περάσαμε σε έναν νέο κύκλο αδύναμης συζήτηση ε, και μείωσης ε, της αύξησης της πίστης. Με τον πληθωρισμό τώρα πολύ χαμηλότερα από τον στόχο μας, η ΕΚΤ αντιμετώπιζε μια νέα πρόκληση. Δεν έπρεπε μόνο να επηρεαστούν τα προβλήματα της νομισματικής ε, μετάδοσης που είχαν δημιουργηθεί από τις τράπεζες οι οποίες απομόχλευαν, αλλά και να επεκτείνουμε την πολιτική μας για να αντισταθμίσουμε τις αποπληθωριστικές πιέσεις. Οπότε τον Ιούνιο του 2014 ξεκινήσαμε τις στοχευμένες μας επιχειρήσεις αναχρηματοδότησης που και πάλι παρήχαν μακροπρόθεσμη ρευστότητα στις τράπεζες υπό τον όρο όμως να δίνουν δάνεια στον ιδιωτικό τομέα. Περάσαμε σε αρνητικά επιτόκια όσον αφορά τα αποθεματικά για να ενθαρρύνουμε περαιτέρω τις τράπεζες να δανείσουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και κατόπιν ανακοινώσαμε το πρόγραμμα αυτό αγοράς περιουσιακών στοιχείων το οποίο αφορούσε αξιόγραφα και ομόλογα και ε, όμως ο πληθωρισμός συνέχιζε να πέφτει τον ε, Ιανουάριο του 2015 επεκτείναμε αυτό το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων για να περιλάβει αξιόγραφα του δημοσίου τομέα. Έκτοτε και η έκταση και η διάρκεια των αγορών μας ε, μεταβλήθηκαν ανάλογα με τις προοπτικές του πληθωρισμού. Επίσης, οι αγορές μας αυτές συμπληρώθηκαν από περαιτέρω μείωση των επιτικίων ε, και της χρήσης αυτού το οποίο λέμε μελλοντικέ κατευθύνσει δηλαδή. Λέγαμε ποιε είναι οι προσδοκίε μα για τη μελλοντική πολιτική μαζί με τι συνθήκε που θα επέφεραν την αλλαγή αυτή. Αυτό συνεισέφερε στη μείωση της αβεβαιότητας σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια, βοηθώντας έτσι να δημιουργηθούν ή να διατηρηθούν οι κατάλληλες χρηματοπιστωτικές συνθήκες. Η στήριξη αυτή κατέληξε σε μια σταθερή ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζώνης. Τώρα έχουμε 22 συνεχόμενα τρίμενα ανάπτυξης. Έχουμε 9,6 εκατομμύρια περισσότερους εργαζόμενους στην Ευρωζώνη από ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2013 που ήταν το χειρότερο σημείο της κρίσης. Σε πέντε χρόνια δηλαδή μέσα το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 7,9% το χαμηλότερο από το 2008 και το ποσοστό απασχόλησης ε, ατόμων 15 ε, μέχρι 74 ετών ανέβηκε από το 54% το 1999 στο 59% στο δεύτερο τρίμηνο του 2018 το υψηλότερο ποσοστό που έχει ποτέ καταγραφεί στην Ευρωζώνη. Ο βασικός κινητήρας της ανάκαμψης είναι η εγχώρια οικονομία. Με μια ενίσχυση της εγχώρια συζήτησης και βελτίωση της αγοράς εργασίας. Αυτή η δυναμική της οικονομίας μας μας κάνει αισιόδοξου πως θα συγκλίνει και ο πληθωρισμός προς τον στόχο μας. Έτσι, από το 2017 και μετά, σταδιακά μειώσαμε το ναι, μηνιαίο ρυθμό αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Αποφασίσαμε πέρσι τον Δεκέμβριο να ολοκληρωθεί αυτό το πρόγραμμα καθώς είμαστε σίγουροι πως η σύγκληση του πληθωρισμού με τον στόχο μας θα συνεχιζόταν. Ταυτόχρονα, οι πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις ήταν πιο αδύναμες από ό,τι περιμέναμε και οι αβεβαιότητες που σχετίζονται κυρίως με παγκόσμιους παράγοντες ε, παραμένουν. Οπότε, δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης. Εξακολουθεί να απαιτείται σημαντικό κομμάτι ε, στήριξης και κινήτρων στην νομισματική πολιτική. Οι μελλοντικέ μας ε, προσδοκίες για τα επιτόκια της ε, ΕΚΤ που ενισχύονται από την επανεπένδυση μεγάλου μέρους των περιουσιακών στοιχείων που έχουμε ήδη αποκτήσει συνεχίζουν να παρέχουν ε, σημαντικό κομμάτι της νομισματικής στήριξης για να διατηρηθεί ο πληθωρισμός κοντά στον στόχο μας. Οπότε τι έχουμε μάθει από την εμπειρία μας. Το νομισματικό μας πλαίσιο βασίζεται σε τρία στοιχεία. Μια σαφή έντολη για να επιτύχουμε σταθερότητα των τιμών. Ανεξαρτησία όσον αφορά τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιτύχουμε την έντολη μας και ένα ισχυρό πλαίσιο λογοδοσίας. Η σημασία του κάθε ενός από αυτά τα στοιχεία ενισχύθηκε από την κρίση. Πρώτα απ' όλα είδαμε ότι μια ξεκάθαρη εντολή έχει μεγάλη σημασία για την αξιοπιστία μας στα μάτια του κοινού. Γιατί εγγυάται ότι η ΕΚΤ θα δρά πάντα για το όφελος ολόκληρης Ευρωζώνης και ε, δεν θα καθορίζεται από ομάδες συμφερόντων. Δεύτερον, η ανεξαρτησία αυτή έχει σημασία σε μια αποτελεσματική νομισματική πολιτική, καθώ επιτρέπει στην Κεντρική Τράπεζα να δρά γρήγορα και ευέλικτα απέναντι σε κραδασμού, ειδικά σε καιρού όπου υπάρχουν δυσκολίε. Ένα, μια λοιπόν εργαλειοθήκη, η οποία θα περιέχει τυπικά και μη μέσα είναι κάτι το οποίο αποδείχτηκε απολύτως απαραίτητο στην περίπτωση στην οποία υπάρχουν προβλήματα στο μηχανισμό νομισματικής μετάδοσης ή δεν υπάρχουν περιθώρια μείωσης των επιτοκίων. Τρίτον, είδαμε την σημασία που έχει το πλαίσιο της λογοδοσίας, ειδικά όταν η Κεντρική Τράπεζα πρέπει να χρησιμοποιήσει νέα μέσα τα οποία δεν είναι εύκολα αντιληπτά από το κοινό. Οι κεντρικές τράπεζες είναι ισχυρές και ανεξάρτητες, αλλά δεν εκλέγονται. Ο συνδυασμός αυτός μπορεί να τετραγωνιστεί μόνο εάν λογοδοτούν σε έρετες αρχές. Έτσι, εντείναμε τις προσπάθειες μας για να βελτιώσουμε την επικοινωνία και την λογοδοσία μας τα τελευταία χρόνια. Το ΔΣ έχει ξεκινήσει να δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων νομισματικής πολιτικής, η ΕΚΤ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ συχνότερα σε επαφή και έτσι έχουμε πολύ περισσότερες ευκαιρίες για να εξηγήσουμε τις αποφάσεις μας και να δείξουμε το πώς δρά η ΕΚΤ σύμφωνα με την εντολή της που είναι ένας βασικός πυλώνας για την νομοποίησή μας. Η κρίση επίσης ε, μας έδωσε αρκετά μαθήματα πέρα από την νομισματική πολιτική. Η Ευρωζώνη μπήκε στην κρίση με ένα ελλειπές θεσμικό πλαίσιο, όχι μόνο για τον τραπεζικό τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς οικονομικής πολιτικής. Η δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας ενίσχυσε τις δυνατότητες των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν την κρίση. Οι μεταρρυθμίσεις στο εθνικό επίπεδο και η πολιτική προσήλωση στο ευρώ που επέδειξαν οι πολιτικοί επίσης έπαιξαν κέριο ρόλο στο κοινό μας εγχείρημα. Αλλά βεβαίως οι αλλαγές αυτές χρειάστηκαν χρόνο, χρόνο ο οποίος χάθηκε από την ανάκαμψη της Ευρωζώνης. Η νομισματική μας ε, ένωση τώρα είναι σε καλύτερη κατάσταση, αλλά πρέπει και μπορεί να σημειωθεί υπεραιτέρω πρόοδος. Όπως είχα την ευκαιρία να πω πριν από την ακρόασή μου στην Επιτροπή Οικονομικών και όπως αναφέρει και το σχέδιο ψηφίσματος, προτεραιότητα τώρα είναι να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της Ευρωζώνης. Έτσι θα ενισχυθεί και η μετάδοση η νομισματική σε μελλοντική ύφεση. Θα μπορεί έτσι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα πολιτικής που θα περιλαμβάνει προληπτικά και διαρθρωτικά μέτρα. Για να καταλήξω λοιπόν, οι πρώτες δύο δεκαετίες της Ευρωζώνης ε, αποτέλεσαν μια εξέλιξη στο πώς διεξάγει νομισματική πολιτική η ΕΚΤ απέναντι σε κάποιες άνευ προηγουμένου απειλές στην σταθερότητα των τιμών προσαρμόσαμε τα μέσα μας για να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο αναφέρει η εντολή μας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό όταν και όποτε απαιτείται σύμφωνα με την εντολή μας όπως αυτή καθορίζεται στις συνθήκες και με ολόκληρη την ανεξαρτησία στα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας όπως ορίζει το νομικό μας πλαίσιο. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι η Ευρωζώνη βγήκε από μια κρίση τόσο σοβαρή που απειλούσε την ύπαρξή της κάποιες στιγμές. Έχουμε βγει από αυτήν κυρίως λόγω της ανθεκτικότητας, της ενέργειας και της επιχειρηματικότητας των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και στην εμπιστοσύνη που έδειξαν στην προσήλωση των ηγετών τους στο ευρώ. Η αντίδρασή μας ε, και η αρχιτεκτονική εντωμεταξύ της ΟΝΕ βοήθησαν να βγει η Ευρωζώνη από την κρίση. Με πολλούς τρόπους έχουμε μια ισχυρότερη νομισματική ένωση σήμερα από ό,τι είχαμε το 2008. Αυτό φαίνεται και στο πόσο δημοφιλές είναι το ευρώ μεταξύ των πολιτών που είναι αυτή τη στιγμή στο υψηλότερο επίπεδο από την εισαγωγή του νομίσματος. Αλλά απαιτείται να γίνουν περισσότερα για να ολοκληρωθεί η ΟΝΕ για να μπορέσει να αντέξει μελλοντικέ κρίσεις για να αποδώσει πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί μόνιμη πολιτική δέσμευση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διάφορους τομείς πολιτικής. Μπορώ λοιπόν εδώ πέρα να επενέσω τον ουσιαστικό ρόλο που έχει παίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα χρόνια της κρίσης και είμαι σίγουρος ότι θα παίξει κέριο ρόλο στην ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η αξιοπιστία της ΕΚΤ βασίζεται στην ανεξαρτησία της και αυτό βασίζεται στην λόγοδοσία της σε σχέση με την έντολή της όπως περιγράφουν οι συνθήκες. Το Κοινοβούλιο με το να ελέγχει την ΕΚΤ παρέχει νόμιμοποίηση στην ανεξαρτησία της και μια από αυτή είναι η τελευταία μου ακρόαση ενώπιον τη Ολομέλεια ω πρόεδρο ε, τη ΕΚΤ. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για το πώ διεξήχθη αυτή η διαδικασία κατά τη διάρκεια τη εντολή μου, για τι επαφέ που είχαμε και για την ευκαιρία που μου δώσατε να εξηγήσω την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. για τα λόγια σας προς το Ευρωκοινοβούλιο. Μέχρι τη λήξη της θητείας σας θα συνεχιστεί η συνεργασία μας. Ακόμη και να αυτή ήταν η τελευταία σας παρέμβαση επί του θέματος του συγκεκριμένου. Θα συνεχίσουμε παρόλα αυτά να συνεργαζόμαστε μέχρι την τελευταία στιγμή. Σας ευχαριστούμε λοιπόν που ήρθατε. Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ντομπρόφσκης. Κύριε Ταγιάννη, κύριε Ντράγκη, συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μάτο, τον εισηγητή, και τα μέλη της Επιτροπής ΕΚΟΝ για τη στήριξή τους. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε. Που βρίσκεται εδώ και ο κύριος Ντράγκη. Και είναι και 20η επέτειος ευρώ. Στα 27 χρόνια το ευρώ απέδειξε ότι είναι ένα τρομερά επιτυχημένο νόμισμα, το οποίο το υποστηρίζουν οι πολίτες τουλάχιστον τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων, που πιστεύουν ότι είναι ένα καλό πράγμα για την Ευρώπη το ευρώ. Η όλη συζήτηση για την Κεντρική Τράπεζα και τι δραστηριότητε τη πέρσι ε, και η εξέταση από το Ευρωκοινοβούλιο αυτών των δραστηριοτήτων είναι θέμα δημοκρατική ε, ε, ε δημοκρατική λογοδοσία. Η Κεντρική Τράπεζα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να διδραματίσει. Και η νομισματική πολιτική τη Κεντρική Τράπεζα, όπω προβλέπεται από τη συνθήκη, είναι ζωτική σημασία για να πετύχουμε τη σταθερότητα των τιμών που χρειάζεται η αγορά. Η ανεξαρτησία και η λογοδοσία είναι αλληλένδετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τι προσπαθίε τη Τράπεζα να ενισχύσει την διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία προ του Ευρωπαίου πολίτε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίση, όπω λέει και η έκθεση, η νομοσματική πολιτική μόνη δεν μπορεί να πετύχει του στόχου τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. Και η οικονομία τη Ευρωζώνη θα πρέπει να συνοδεύεται από φιλοδο... φιλόδοξε, στραμμένε προ την ανάπτυξη κοινωνικά ε, εύρωστε δημοσιονομικέ πολιτικέ βάση και με το Σύμφωνο ε, Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να επιταχύνουμε την αγορά ε, την, την ένωση των κεφαλαίων για να έχουμε ανθεκτικότητα σε διάφορους τριγμούς και κλειδονισμούς ε, ώστε να ενισχυθεί και η νομισματική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη της έκθεσης ότι η Ένωση των Κεφαλαγορών με την ε, βήμα-βήμα επίσης ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα βελτιώσει την κατάσταση για όλη την Ευρώπη. Το τονίζουμε και στην ανακοίνωσή μα για έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ, όπω υποβλήθηκε στι 5 Δεκεμβρίου πέρσι. Είμαστε βέβαια για την επικοδημοτική συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην όλη διαδικασία και βεβαίω το είδαμε και προηγουμένω με την όλη στάση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα περασμένα χρόνια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Ντελάνγκη για ένα μισή λεπτό. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Μάτο για την πολύ καλή έκθεση του και τον Πρόεδρο της ε, ΕΚΤ ε, για τις γενικότερα θετικές τάσεις που περιγράφονται άλλωστε και στην έκθεση. Διαπιστώνω πως ε, πάρα πολλές τράπεζες χρησιμοποίησαν τον χρόνο αυτό για να εξηγιάνουν τον ισολογισμό τους και πράγματι έχει πέσει το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αλλά υπάρχουν δυστυχώς και εξαιρέσει και είμαι υπερήφανη για το ότι μαζί με τον συνάδελφο Γκουαλτιέρη και ένα πολύ επικοδομητικό και συνεργάσιμο συμβούλιο εργαζόμαστε για να καταρτήσουμε πρώτον κανόνες που θα υποχρεώνουν όλες τις τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουν επιτέλους το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Επιτέλους θα έλεγα. Και βεβαίω αυτό αφορά και τα υφιστάμενα κόκκινα δανεία. Τώρα, για την ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσεων που επίσης ε, είναι θέμα της ε, έκθεση του συναδελφού Μάτο. Νομίζω πως η Μπάνκα Ρέτζιο στην ε, Ιταλία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Γιατί εκεί πέρα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η χρηματοδότηση και η παρέμβαση αυτή για να κεφαλαιοποιηθεί η τράπεζα. Και βεβαίως είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται, αλλά βλέπουμε ότι πάει ο ε, λογαριασμός πάλι στον φορολογούμενο, κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει. Αυτό δείχνει γιατί κάποιες χώρες ε, δεν έχουν ιδιαίτερη όρεξη για ένα ευρωπαϊκό σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Και γιατί να κάνουν κάτι τέτοιο όταν υπάρχουν εθνικά τέτοια. Ε, θεωρώ όμως ότι πρέπει να φύγουμε από αυτήν την συζήτηση γιατί καλύτερη θα ήταν μια λύση στην Ευρώπη και όχι ένα μπλοκάρισμα. Και βεβαίως η πρώτη ευθύνη βρίσκεται στα εθνικά συστήματα εγγύησης καταθέσεων και μετά βεβαίως μπορεί να υπάρξει προσφυγή στο ευρωπαϊκό σύστημα. Έχω μια συγκεκριμένη βεβαίως ε, ερώτηση προς τον ε, κύριο Πρόεδρο, ο οποίος πάντα ήταν υπέρ ενός ευρωπαϊκού συστήματος, θέλετε να ξεκινήσουμε τώρα ή πώς θα περιμένετε την επόμενη θητεία του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μόργανο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον Πρόεδρο Ντράγκη που ήρθε εδώ σήμερα και τον εισηγητή, τον κύριο Μάτο, για την θετική μας συνεργασία ε, στην Επιτροπή ε, ΕΚΟΝ. Χωρίς να επεκταθώ στις λεπτομέρειες της έκθεσης, θέλω να τονίσω την σημασία τη συζήτηση τη έκθεση αυτή και τη έγκρισή τη ιδίω αυτέ τι μέρε που γιορτάζουμε την 20η επέτειο υιοθέτηση του ευρώ. Είναι σκόπιμο να γίνει αυτό τώρα. Γιατί τώρα αντιμετωπίζουμε θέματα χωρίς ε, ανεπανάληπτα στο παρελθόν, διότι το ευρώ είναι ε, ένα μεγάλο κατόρθωμα της ευρωπαϊκής οικοδόμησης, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση στα οικονομικά θεματα χωρί ε είναι ακόμη ολοκληρωμένη. μεγαλο κατορθωμα τη Ευρωπαϊκή οικοδόμηση, αλλα η κοινωνική ειναι ακομα ολοκληρωμενη λειπουν λειπει η φορολογική διάσταση, Έχουμε τις πιο ορατές αδυναμίες ε, εδώ ε, και όταν ακούν αυτές τις αξιολογήσεις οι πολίτες ε, πραγματικά τους ενδιαφέρει. Η λιτότητα δεν μπορεί να είναι η μόνη μα απάντηση. Η αλληλεγγύη και η ευθύνη είναι η μόνη κατάλληλη αντίδραση. Πρέπει λοιπόν να αναλυθούν εθνικέ πρωτοβουλίε για το ευρώ. Κάθε φορά ορίζονται από το κεντρικό επίπεδο περαιτέρω βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν και η συνέπεια είναι ότι 20 ε, χρόνια μετά τη δημιουργία του ευρώ συζητάμε το τεχνοκρατικό επίπεδο του έντις και το τι θα γίνει με τα κοινωνικά δικαιώματα και πάβο. Εδώ ε, θα πρέπει η συζήτηση για την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να ασχοληθεί ε, με αυτό που ε, με, άριστο τρόπο καταφέρατε και εσείς κύριε Ντράγκη προεδρεύοντας εκεί. Εδώ οι ευρωβουλευτές ε, θα πρέπει να δούμε υπό το φως και των πρόσφατων συμπερασμάτων του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου το όλο θέμα. Τα έκτακτα μέτρα της νομοσματικής πολιτικής που υιοθέτησε και η ε, Κεντρική Τράπεζα είναι απαραίτητα για την Ευρωζώνη, αλλά οι πολίτε μα έχουν υποφέρει και από την κρίση. Θα πρέπει λοιπόν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα προστασία. Τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε συνεπεί μεταξύ των όσων λέμε και των όσων πράττουμε. Και όχι να περιχαρακωνόμαστε σε εθνικά οχυρά. Ευχαριστούμε, Πάκετ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κύριε Ντράγκη. Πριν από 10 χρόνια ξέσπασε η οικονομική κρίση, η οποία ξέφυγε στην Ευρώπη γιατί υπήρχε πάρα πολύ χρέος και πολύ φθηνό χρήμα. Και ποια είναι η απάντηση της ΕΚΤ, ακόμα περισσότερο χρέος και ακόμη φθηνότερο χρήμα. Οπότε διαβάζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε εδώ πέρα στην έκθεση, το οποίο έχει όμως σοβαρές συνέπειες. Οι και οι συντάξεις έχουν προβλήματα. Οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται τεράστια. Δεν μπορεί ο απλός άνθρωπος να αγοράσει πλέον ακίνητα. Έχουμε επίσης αύξηση του χρέους των επιχειρήσεων, των οικοκυριών και κυρίως των κρατών. Και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, ειδικά στις χώρες που τις χρειάζονται περισσότερο, αναβάλλονται συνεχώς. Και πλέον είναι τόσο χαμηλά τα επιτόκια, ώστε καταδικάζονται οι αποταμιευτέ. Ο απλός άνθρωπος στον δρόμο. Ένας άνθρωπος στην ηλικία μου που δεν είχε ούτε μία σχέση με το θέμα όταν ξεκίνησε η κρίση το 2018 πραγματικά απελπίζεται από την πολιτική τραπεζών και κρατών. Είμαστε στο τέλος εντολή σα. Επί χρόνια μας λέγατε πως είστε ο πυροσβέστης που έζησε τη φωτιά. Φοβάμαι όμως ότι η πολιτική αυτή μοιάζει με πολιτική ενός πυρομανούς που θα οδηγήσει στην επόμενη οικονομική κρίση. Σας ευχαριστώ. Αρτουή για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, κύριε Σεγητά, συνάδελφοι. Τη στιγμή που η θητεία μας οδεύει προς το τέλος της, θα πρέπει να αποφανθούμε για την έκθεση αυτή, την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ε, και λόγω της περίστασης αυτής της 20ης επαιτίου υιοθέτησης του ευρώ είμαστε και συγκινημένοι κύριε Ντράγκη. Είναι η τελευταία σας παρουσίαση και παρέμβαση εδώ ενώπιον αυτής της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου. Τα μηνύματα τη έκθεση αυτή είναι πολλαπλά. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ε, φέρει ει πέρα περισσότερο από ε, ορθότατα την αποστολή που ανέλαβε. Και ενώ τα προβλήματα είναι ατελείωτα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βέβαια δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πρέπει και τα κράτη-μέλη να επαγρυπνούν για τι δημόσιε δαπάνε του, για τον έλεγχο των δημοσιονομικών του και για την ε, ε, καλή διαχείριση των οικονομικών του προ όφελο των πολιτών και των ευρωπαϊκών στόχων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα θα επαγρυπνεί και εκείνη για τα διάφορα προβλήματα, όπω τι τιμέ ε, στην αγορά κινήτων ή την τα δάνεια που ε, πρέπει να παρακολουθεί με προσοχή και τις μελλοντικέ επενδύσεις. Νομίζω ότι η αναγνωρισμένη επιτυχία του ευρώ είναι πραγματικά κάτι το αξιοθαύμαστο. Διότι πριν από 20 χρόνια είχαμε μια ε, ε, τη γένεση ενός νομίσματος χωρίς να τα, είναι προσδεδεμένο σε κάποιο συγκεκριμένο κράτος. Και έτσι θα πρέπει σύντομα να προβλέψουμε για την Ευρωζώνη την απαραίτητη οικονομική, δημοσιονομική, φορολογική, τραπεζική και κοινωνική διακυβέρνηση ώστε να ε, επουλώσουμε, να θεραπεύσουμε αυτή την αρχική της αναπηρία. Θα πρέπει να δούμε τις παγκόσμιες πιέσεις που δεχόμαστε και να αντιδράσουμε. Θα πρέπει το ευρώ να γίνει ένα όπλο, όπως έχουν κάνει, είπαμε, το δολάριο. Θα πρέπει να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ε, τις καταστάσει όπου θα πρέπει να επιβληθούν και ποινέ ή πρόστιμα σε τράπεζε ή θεσμού τρίτων χωρών. Θα πρέπει λοιπόν να αναγνωρίσουμε πόσο το ευρώ ε, βοηθά στην ανθεκτικότητα και αντοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Η προστιμα σε τραπεζε η θεσμου τριτων χωρων θα πρεπει λοιπον να αναγνωρισουμε ποσο το ευρω βοηθα στην ανθεκτικοτητα και αντοχη τη ευρωπαικη ενωσης η κεντρικη τραπεζα και το ευρώ είναι σύμβολα τη εμπιστοσύνη μα στο μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω προσοχή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν πρέπει να είναι δεκανίκη τη ε, ε, ε, πλημελού πολιτική διαχείριση. Ευχαριστούμε κύριε Σορτασούν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τα μη συμβατικά μέτρα διατήρησε την Ευρωζώνη σε κατάσταση επίπλευσης, όμως πρέπει να δούμε κάποια στοιχεία εκδημοκρατισμού και ξέρετε μας ανησυχεί ε, η αγορά περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τον άνθρακα δεν συνεισφέρουν ε, στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όμως αυτό που θέλουμε να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που ξέρουμε ότι χρειάζεται η Ευρωζώνη για να αποφύγουμε μελλοντικέ κρίσεις και μας ανησυχεί ότι ένας είναι συνοψισμός μεταξύ αυτών που ε, δεν θέλουν να μειώσουν τους κινδύνους και κάποιων που θέλουν να τους αμοιβεοποιήσουν να υλοποιείται. Ε, δηλαδή πρέπει να έχουμε έναν προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, διαφορετικά οι αδυναμίες θα είναι πολύ μεγάλες και σίγουρα πρέπει να κάνει αυτό το άλμα ε, το ευρώ μετά από 20 χρόνια από τη δημιουργία του. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Κάθη για ένα λεπτό. Κάρθη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ε, ε, έχει προστατεύσει τα κράτη-μέλη και τι τράπεζέ του από τι πιέσει που δέχονται. Σε πολλά κράτη-μέλη, οι κεντρικέ τράπεζε έχουν αποτύχει με τη σειρά του να ε, αποφύγουν τις εξώσει και τις εξαγορές σπιτιών την πώληση μάλλον σπιτιών. Ε, σύντομα θα πολλαπλασιαστεί το φαινόμενο αυτό, θα δεγκωθεί και στην Ιρλανδία. Ε, Πολλέ φορέ ε, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα μπορούσε να είναι ευκαιρία για ισχυρότερη προστασία για του ε, δανειστέ. Ε, Όμω, η προσέγγιση τη Επιτροπή και του Συμβουλίου δείχνουν ότι το μόνο του ενδιαφέρον είναι να ε, φέρουν μαζικό κέρδο στι Ευρωπαϊκέ Τράπεζε. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι δευτερογενεί αγορέ για τα MPL είναι κάτι που θα έχει για μένα θλιβερέ συνέπειε στα δάνεια κινήτων. Θα πρέπει η ΕΚΤ να αρχίσει να προστατεύει από αυτά τα όρνεα του απλού ανθρώπου. Διότι εάν η Κεντρική Τράπεζα και το Συμβούλιο δεν δράσουν, οι πολίτε ρωτάνε ποιοι θα το κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πατήσει πόδι εδώ. Και ε, το Ευρωκοινοβούλιο το ίδιο μαζί με την κοινωνία των πολιτών για να μπλοκάρει αυτή την τάση. Ευχαριστούμε Μόιτα για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Κεντρικής Τραπεζάς, ο απολογισμός σας δεν είναι θετικός. Ε, κάνατε κάποιες ε, προβλέψεις ήδη που αποδείχθηκαν λάθος. Τα επιτόκια είναι σε ιστορικό χαμηλό. Δεν τα έχετε αυξήσει καμία φορά σε 7 ολόκληρα χρόνια. Η Γερμανία, ο κινητήρα τη Ευρωζώνης, είναι στα όρια της ύφεση. Δεν έχετε πλέον καμία άλλη δυνατότητα μείωση των επιτοκίων. Έχετε αγοράσει πάρα πολλά ομόλογα και επεκτείνει κατά πολύ, ορίστε, τον ισολογισμό ε, Τη κεντρική Τράπεζας. Κάνατε του στοχούς στοχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. Ακολουθήσατε την πιο επεκτατική πολιτική που υπήρξε ποτέ. Και έχετε πάρα πολλά ομολόγα και της Γερμανίας στον ισολογισμό σας. Το θέμα είναι λοιπόν τι θα αφήσετε στους διαδόχους σας. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αναγνωρίσουν ότι είστε υπεύθυνος για την οικονομική καταστροφή της Ευρώπης και θα αποκαλυφθεί μια μέρα αυτό. Σας ευχαριστώ. Τζάνι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε Ντράγκη, σήμερα γιορτάσαμε την 20η επέτειο από την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος του ευρώ. Νομίζω ότι είναι καλή συγκυρία για να κάνουμε μια καλή αποτίμηση και το τι έκανε η Ευρωπαϊκή Τραγική Τράπεζα δεδομένων των ε, αριθμών και των συνθήκων στους οποίους ζουν οι πολίτες της Ευρωζώνης. Διότι όλα αυτά ε, τη αξιολόγηση βάσει των δεδομένων δεν τα βλέπω τόσο θετικά. Οι προσχέσεις που δόθηκαν στους Ευρωπαίους πολίτες ιδίω από τη στιγμή της γέννησης του ευρώ και μετά, δεν έχουν πληρωθεί. Το ευρώ έχει φέρει σοβαρότατες ε, αποκλήσεις στο εισόδημα των χωρών. Χαμηλότατη ανάπτυξη σε κάποιες χώρες. Η Ευρωζώνη σήμερα γίνεται αυτό το άθροισμα κρατών, αυτή η ομάδα που αναπτύσσεται λιγότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Η ενεργεία είναι ψηλότατη. Σήμερα έχει διπλασιαστεί σε σχέση με τρίτα κράτη. Και ε, η θητεία σα ω Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν σα επέτρεψε να πετύχετε τα απλώ τα καταστατικά καθήκοντα και στόχου που είδατε. Δηλαδή, δεν υπάρχει ανάπτυξη ούτε αυτόνομη βιωσιμότητα των ποσοστών που είχαμε ορίσει. Έχει ε, δαπανηθεί ένα πακτολό χρημάτων και κονδυλίων που δεν έχουν φτάσει στην πραγματική οικονομία. 29 μόνο ε, έφτασαν, ε, από τα δίσκη που ξοδεύτηκαν έφτασαν σε οικογένειε που τα χρειάζονταν. Εδώ λοιπόν λίγα νομίζω είναι αυτά για τα οποία θα πρέπει να γιορτάσουμε. Και είναι μια στιγμα... σημαντική στιγμή περισυλλογή για όλου μα για να δούμε γιατί απέτυχε το ευρώ και ιδίω εσεί ω διευθυντή τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη θητεία σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Ζαριανόπουλο για ένα λεπτό. Παρά τι συναυολογίε για την ευρωενωσιακή οικονομία, π.χ. την δίθε μείωση τη ανεργία με γεννή και τη ημερική απασχόληση, δεν μπορείτε να κρύψετε του φόβου σα. Ανεμική ανάπτυξη, επιβράδυση, ανισομετρία, προστατευτισμοί, εμπορικοί πόλεμοι που πολλέ φορέ γίνονται θερμοί με χιλιάδε θύματα, Brexit, πολιτική αναταραχή και φόβο νέα χειρότερη κρίση. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο καπιταλισμό. Κάνετε συστάσει απειλέ, συνέχιση αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων φοροαπαλλαγέ στο κεφάλαιο φοροκυνηγητό στο λαό μισθοί κατά την προαίρεση και τα κέρδη των καπιταλιστών κατάργηση συλλογικών συμβάσεων επιβίωση με επιδόματα ψίχουλα και οι τράπεζε που ελέγχεται με απολύσει παράδειγμα στην ελλάδα δεκαπέντε χιλιάδων τουλάχιστον τραπεζοϊπαλλήλων την επόμενη διετία χιλιάδε πληστηριασμοί θηλιά στο λαιμό εκατομμυρίων ανθρώπων ή ρυθμίσει με το πιστόλι στον κρόταφο για κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και των κερδοσκοπικών funds μνημόνια δηλαδή γενικευμένα και διαρκεία το ψευτοδήλημα συντήρηση πρόοδο πάει να κρύψει την ενιαία στρατηγική σύμπλευση ακροδεξιά συντηρητικών σοσιαλδημοκρατών νεοαριστερών τύπου τσίπρα που συγχαίρουν Μέλκερ και τραμπ. η διαφορά είναι στην οργανωμένη του λαού στην ενίσχυση των κομμουνιστών για την ανατροπή αυτής τη βαρβαρότητας. Κύριε για την 20η ε, επέτειο του ευρώ και την ε, επέτειο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής ε, Τράπεζας πριν λίγους μήνες. Σε αντίθεση με άλλους ομιλητές είμαι επιβεβαισμένος ότι μπορείτε να είστε περήφανος για το πώς ασκήσατε τα καθήκοντά σας. Ήσασταν πολύ αποτελεσματικό στο να αντιμετωπίσετε την υπαρξιακή κρίση τη Ευρωζώνη το 2012 και χάρη στην αποφασιστική σα τάση νομίζω ότι επιβίωσε το ευρώ και τώρα ανθίζει. Πολλές από τις επικρίσεις που ακούσαμε πριν λίγα λεπτά απλώς μας δίνουν μία εικόνα άγνοιας από την πλευρά κάποιων συναδέλφων. Δυστυχώς δεν καταλαβαίνουν πώς εργάζεται, πώς λειτουργεί η νομισματική πολιτική. Αυτά για το παρελθόν τώρα, για το μέλλον. Νομίζω εμείς και η ΕΚΤ αντιμετωπίζει τρεις κυρίες προκλήσεις. Θα πρέπει να δούμε ότι η ύφεση ε, συμβαίνει στην ευρωπαϊκή οικονομία και μάλλον θα έχουμε μια ακόμα κρίση. Είναι έτοιμη η να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση. Νομίζω το σημαντικό είναι ότι πρέπει να έχετε περιθώριο ελιγμών στην νομισματική πολιτική γιατί το μηδενικό ποσοστό επιτοκίων δεν δίνει μεγάλη ευελιξία από τη σκοπιά της νομισματικής πολιτικής για να βοηθηθεί η οικονομία. Και τέλο, το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό ταμέα πρέπει να επιληθεί γρηγορότατα. Σας ευχαριστούμε. κυρία Μπρέσο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τον κύριο Ντράκη για το έργο τους σήμερα. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του ευρώ και αυτή η έκθεση μας υπενθυμίζει επίσης το σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Κεντρική Τράπεζα τα τελευταία χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κοινό νομισμά σε μια τόσο δύσκολη στιγμή αποτελεί σημαντικό μήνυμα η ε, διατήρηση της νομισματικής ε, πολιτικής της Ένωσης και στην ανάπτυξη της ε, Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Όμως ήταν σημαντικό η ΕΚΤ να λάβει υπόψη και τις κοινωνικές συνέπειες των πολιτικών της, όπως ζητείται από τη Συμφωνία των Παρισίων. Η πρόσφατη περίπτωση με την τράπεζα Κάριτσεμ στην Ιταλία μας δείχνει ένα θετικό ρόλο που μπορεί να παίξει η την στην προστασία των μικρών επενδυτών ε, και αποταμιευτών. Πρέπει να γενικεύσουμε αυτό το ρόλο ε, προωθώντας την ε, λογική της συμπλήρωσης και υλοποίησης της Τραπεζικής Ένωσης και με ένα σύστημα ασφάλισης των καταθέσεων. Ε, εμείς ε, περιμένουμε μελλοντική πρόοδο και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία για το τέλος της θητείας σας. Ο κύριος Λούκε, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, το Κοινοβούλιο γιορτάζει σήμερα τα 20 χρόνια του ευρώ, αλλά τι γιορτάζουμε τελικά. Δηλαδή αν είμαστε ειλικρινεί, πρέπει να πούμε ότι το ευρώ μας έχει φέρει τη μία δυσκολία μετά την άλλη. Ας δούμε παραδείγματος χάρη την κρίση του δημοσίου χρέους. Ποτέ δεν είχαμε, δεν θα είχαμε τέτοια κρίση εάν δεν είχαμε το ευρώ. Γιατί βεβαίως τα κράτη που έχουν εθνικό νόμισμα μπορούν να αναχρηματοδοτούν το χρέος τους, τυπώνοντας. Και βεβαίως δεν θα είχαμε την παγκόσμια κρίση σε αυτήν την έκταση χωρίς το ευρώ. Και βεβαίως ε, βρέθηκαν τελικά οι τράπεζες να έχουν τεράστια ε, ποσά σε κρατικά ομόλογα, τα οποία μετά τα κράτη βρέθηκαν σε δυσκολία να εξυπηρετήσουν, γιατί όπως είπαμε δεν μπορούσαν να τυπώσουν χρήμα. Στην ε, Νότια Ευρώπη τεράστια ανεργία των νέων. Όλα αυτά οφείλονται στο ευρώ. Δεν έχουμε τίποτα να γιορτάσουμε λοιπόν. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε κάπως αυτά τα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύτηκαν. Το ευρώ είναι ένα τελείως αποτυχημένο πείραμα. Σας ευχαριστώ. Πεντιτσίνη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Ντράγκη, εγώ σας μιλώ ως Ιταλός, δηλαδή ως πολίτης μιας ε, χώρας που ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι η τρίτη χώρα μεταξύ των ε, εισφερόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 25 χρόνια σημειώνει πρώτη δηλαδή έχουμε Ιταλούς που έζησαν πάνω από τις ε, δυνατότητές τους ε, και ε, μόνο χάρη στους τόκους ενός χρέους που έχει αυξηθεί ανάλογα χάρη στη δεκαετία του 80 και χάρη σε επιτόκια 10% πραγματική καταστροφή. Φτάσαμε λοιπόν στα 2.300 δημοσίου χρέους και ε, έχει πληρώσει τεράστιους ε, τόκους η Ιταλία, δηλαδή ε, έχουν ξεπεράσει οι τόκοι το ίδιο το χρέος και τώρα το αγοράζουν το χρέος οι τράπεζες της Γαλλίας και της Γερμανίας, αλλά ακόμη και έκτισε με πολύ χαμηλά επιτόκια χωρίς κανένα όρο και οι τράπεζες μπόρεσαν λοιπόν να κερδοσκοπήσουν και δυστυχώς το αγοράζουν και με χρήματα που έχουν δημιουργηθεί από το πουθενά. Βάζουν απλώς μηδενικά στους υπολογιστές και αυτούς τους τόκους τους πληρώνουν οι Ιταλοί με την πραγματική οικονομία, με τον πραγματικό τους υδρότα, όχι με έναν υδρότα που προέρχεται από το πουθενά. Όμως φαίνεται αυτό το σύστημα να τους ικανοποιεί όλους, οι τράπεζες είναι ικανοποιημένες ε, γιατί ε, τελικά... Ε, ε, επανισάγουν ε, τα δικά τους κεφάλαια ε, και δυστυχώς πληρώνει η πραγματική οικονομία. Είναι οι μικρές και μεσές επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση στην πίστοση. Και φυσικά έχουμε και αύξηση της ανεργίας. Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε σε τρομακτικά νούμερα στις χώρες όπου είχαμε αύξηση δημοσίου χρέους, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία δυστυχώς. Έχουμε το άρθρο 127 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου λέγεται ότι πέρα από τη σταθερότητα των ε, τιμών, είπατε εσείς ότι το πέτυχε αυτό, η ΕΚΤ ε, θα πρέπει να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά πολέμηση ενεργείας και προώθηση ισορροπημένης οικονομικής ανάπτυξης. Η ερώτησή μου είναι, η ΕΚΤ έχει πράγματι σκοπό να καταπολεμήσει την χρηματοοικονομική κερδοσκοπία και να δράσει με ένα διαφοροποιημένο τρόπο για ε, να μειώσει τα σπρέτ των μερμένων κρατών ε, μελών ε, και μπορεί να επιδράσει στο μηχανισμό το σπρέτ που καταστρέφει η οικονομία κρατών όπως στην Ιταλία και αποδυναμώνει ή καταστρέφει και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Πρέτσελ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ντράγκη, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του ευρώ, αλλά γεγονός είναι πως οι ανισορροπίες εντός της ευρωζώνης εξακολουθούν να είναι τεράστιες. Αυτό φαίνεται βεβαίως ε, και στο χρέος και στην εξέλιξη τη βιομηχανική στη Γαλλία και στην ε, Ιταλία φαίνεται επίσης ε, και στην εξέλιξη των μισθών στην Γερμανία η Ευρωζώνη ανήκει στις ε, περιοχές εκείνες ε, με την χαμηλότερη οικονομική ανάπτυξη στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Έχουμε κομμάτια της Αφρικής που τα πάνε πολύ καλύτερα τα τελευταία χρόνια από ό,τι Ευρωζώνη. Ίσως η Βενεζουέλα να τα πηγαίνει χειρότερα, όπως ισχύει άλλωστε σε όλες τις σοσιαλιστικές χώρες. Γεγονός είναι πως αυξάνονται τα κρατικά χρέη και είστε συνυπεύθυνος εσείς κύριε Ντράγκη. Σας ευχαριστώ κύριο Συναδεινός για να λεπτό. Κύριε Ντράγκη, πίσω από τη δική σας θεσμική υπόσταση, πραγματική υπέτειη σε αυτό το θέατρο σκιών είναι η εντολή σας και όσοι εθνικοί ηγέτες που παραδομένοι στις υποσχέσεις το εφήμερο όφελος και το παροδικά φθηνό χρήμα παρέδωσαν κυριαρχικά δικαιώματα υποθήκευσαν την περιουσία των πολιτών και ξεπούλησαν εθνικές αποταμιεύσεις είστε ένας κεντρικός τραπεζίτης που ελέγχει την προσφορά του χρήματος αλλά δεν εντέλεται την τόνωση της ζήτησης υπεύθυνος για τη σταθερότητα των τιμών αλλά όχι για την ευρωστία της οικονομίας τη μεγιστοποίηση υγιούς εργασιακής απασχόλησης και της ενίσχυσης των μισθών και της αγοραστικής δύναμης. προσφέρατε τα πάντα για μια ένωση κατ' επιταγή και με αποκλειστικό όφελος της γερμανίας και των δορυφόρων της για μια γερμανία που από το 2008 εξοικονόμησε χάρη στα δικά σα χαμηλά επιτόκια δανεισμού 368 δισεκατομμύρια ευρώ. κάθε σα πράξη αποδεικνύει τι στρεβλώσεις του οικοδομήματος ένεκα πολιτικών και μεροληπτικών αποφάσεων. μια κεντρική τράπεζα μιας ατελούς ένωσης με περιορισμένες ευθύνε και λήψη εντολών. ευχαριστώ. <clears throat> Uh, Ευχαριστούμε. Κεντελάρα για Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Έχουμε σήμερα την 20η επέτειο του ευρώ, αλλά πριν από λίγα χρόνια πραγματικά είχαμε ε, την απορία για το εάν θα επιζήσει το ευρώ. Γιατί λοιπόν ήταν ε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αυτή η οποία εκλήθη να αντιμετωπίσει αυτήν την ε, κρίση. Πρώτα απ' όλα, όταν, όταν φτιάχτηκε το ευρώ, Πρώτα υπάρχει μια πολιτική ολοκλήρωση και μετά ακολουθεί το νόμισμα. Στην περίπτωσή μας έγινε το αντίστροφο και μας είπαν τώρα σκάσε και κολύμπα. Έχουμε λοιπόν τεράστιες οικονομικές ε, διαφορές οι οποίες δεν μπορούν να γεφυρωθούν μεταξύ των κρατών ε, μελών ε, γιατί δεν υπάρχουν και οι απαραίτητοι μηχανισμοί αλληλεγγύης. Γιατί λοιπόν έπρεπε να σώσει η ε, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ευρώ. Λόγω της ε, ίδιας του της ε, φύσης, ε, λόγω της οικοδόμησης του. Σήμερα λοιπόν έχουμε προχωρήσει παρακάτω, αλλά είτε θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, είτε θα ξαναγίνουν τα ίδια πράγματα και προσεχώς. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νόμισμα το οποίο θα έχει επαρκούς, επαρκείς μηχανισμούς αλληλεγγύης και θα βοηθήσει και τις ε, τράπεζες και τις χρηματοφορές. Σας ευχαριστώ. Ρούνεν για ένα λεπτό. Οι ευρωπαϊκές η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη έκθεσή τη λέει πω το 2018 αναπτύχθηκε γρηγότερα από ποτέ η ευρωπαϊκή οικονομία.